Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Κυρίσω την επανάληψη ε, της Συνόδου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπτει στις 13 ε, Σεπτεμβρίου 2012. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Έχετε αντιρρήσεις.